Κυρίες και κύριοι, η Σύνοδος θα συνεχιστεί αύριο, 5η 16, ε, 3η 16 Απριλίου 2013, από τις 9 μέχρι τις 2 και από τις 3 μέχρι τις 11 το βράδυ.